Ζανώνη υπό την προπόθεση ότι δεν καταλαμβάνει κάποιο αξίμα που δεν συνέβη με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλο, έλαβα από τον κύριο Λουίτζι Νταματζίστη, ε, πρώην ε, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα αίτημα υπεράσπισης ε, της κοινοβουλευτικής του ασυλίας ε, και προνομίων ε, στα πλαίσια μιας δικαστικής αγωγής στο Λαμέτσια Τέρμε. Πρόκειται για ένα πρωτοδικείο στο Λαμέτσια Τέρμε και βάσει το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού θα αναπέμψουμε το αίτημα αυτό στην καθήλια αρμόδια επιτροπή. Και τέλος... Βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 4 του ιστορικού κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 11 Ιουλίου του 2011 επαλή